Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να καταδείξουμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ε, ημερήσιας διάταξης. Τα άμεσα μέτρα της Ένωσης για την στήριξη της Ιταλίας και των άλλων κρατών μελών που επηρεάζονται από έκτακτη συρροή μεταναστών. Δίνω το λόγο στην Επίτροπο, την κυρία Μάλστρον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, σα ευχαριστώ για αυτή την εξαιρετικά επίκαιρη συζήτηση. Οφείλουμε ε, να εξετάσουμε την τωρινή κατάσταση. Η Επιτροπή την παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ. Ο Frontex έχει στείλει δύο επί επιτόπου. Περίπου 5.500 μετανάστε από την Τινησία έχουν φτάσει στι Ιταλικέ ακτέ ε, τι τελευταίε ημέρε. Ε, και έχουν τροποποιηθεί τα τελευταία 24 ώρο κατά τι αυτά τα νούμερα. Όσοι καταφθάνουν είναι κυρίως άντρες, ε, γύρω στα 30 χρόνια, ε, υπάρχουν όμως και 30 γυναίκες και 108 παιδιά. οι 27 διευκολυντέ εντοπίστηκαν, παράνομοι διευκολυντέ. Έφτασαν λοιπόν οι τηρήσει οι μετανάστες στις Ιταλικές ακτές και προφανώ πιέζουν το κέντρο υποδοχή στη Λαμπεντούζα. Ήδη το περασμένο Σάββατο ήρθαμε σε επαφέ με το Υπουργείο Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας. Επίσης, λάβαμε μία επιστολή, μία επίσημη αίτηση για την χορήγηση βοήθειας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να βοηθήσουμε και την Ιταλία και την Τινησία. Είναι ένα θέμα, όχι διμερές, είναι ένα θέμα που αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και πριν τις τελευταίες εξελίξεις, η, Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγγνώμη, και ο Frontex ε, ε, προσπάθησαν να εξετάσουν την μεσομακροπρόθεσμη πολιτική. Όλα θα πρέπει να εδράζονται επί της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ήδη συνδράμουμε την Ιταλία. Η προσέγγιση προσέγγιση μα επίση θα πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη με την Τινησία για να τη στηρίξουμε στη δημοκρατική ε, μεταβατική αυτή, συγγνώμη, στην μεταβατική αυτή περίοδο. Και αυτό είπε σήμερα η κυρία Άστον στην Τινησία. Προσέφερε δε και υλικοτεχνική και οικονομική στήριξη. Ε, των συνθήκων έχουμε ε, εντοπίσει συγκεκριμένα μέτρα αλλά και ταχεία οικονομική βοήθεια. Από οικονομική ε, πλευρά θα χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Μεταναστών για το 2011, πέρα από τη χρηματοδότηση που ούτω ή άλλω σκοπεύαμε να αφιερώσουμε στην Ιταλία. Ε, υποδομές, υλικοτεχνική στήριξη, ιατρική βοήθεια, κοινωνική βοήθεια, ε, σύμβουλοι, διοικητική βοήθεια με τις διαδικασίες ασύλου, γλωσσική βοήθεια, είναι στοιχεία που περιέχονται στην αρρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης θα κινητοποιηθεί και το Ταμείο Συνόρων και η Ιταλία μπορεί να απευθυνθεί και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων τη Λαβαλέτα για να επιτύχει μεγαλύτερη υποστήριξη προς τις εθνικές αρμόδιες αρχές που ασχολούνται με τα θέματα ασύλου. Μη, ε, θα μπορούσαμε επίσης να οργανώσουμε μια κοινή ε, επιχείρηση Frontex. Είμαστε σε στενή επαφή με το Frontex και προετοιμαζόμαστε σε τεχνικό επίπεδο. Ως συνήθως ε, αυτή, ε, το αποτέλεσμα θα βασιστεί ε, στην συνδρομή των κρατών μελών ω προ τον εξοπλισμό και ζητώ τη βοήθειά σα, ζητώ την στήριξή σα. Θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω όμω για το εξή σε σχέση με τη συζήτηση που μόλι ολοκληρώθηκε. Επειδή είναι διαφορετική φύση οι χερσαίε και οι θαλάσσιε επιχειρήσει ε, και επειδή κάποια νέα κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν στην κοινή επιχείρηση, α μην ξεχνούμε ότι έχουμε και στην ελληνική μεθόριο μια προϊούσα επιχείρηση που επίση στα προτεραιότητα. Επίσης ε, υπάρχουν ευπαθεί ε, πληθυσμιακέ ομάδε άλλοι που χρήζουν διεθνού ε, προστασία. Όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και να εξασφαλιστεί η ειδική προστασία για όσους το χρειάζονται όπω προβλέπεται από το κοινοτικό και από το διεθνέ δίκαιο και για τι μεμονωμένε δράσει. μπορώ να σα πω ότι είμαστε έτοιμοι να συσκεφθούμε με τι ιταλικέ αρχέ για να αποφασίσουμε για τι λεπτομέρειε του σχεδίου δράση και τα επόμενα βήματα. Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, Φυσικά πρέπει να εκπονήσουμε και μία μεσοπρόθεσμη στρατηγική, κυρίω για τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική διαχείριση των συνορών αλλά και στρατηγική για να υποστηρίξουμε τη δημοκρατική μετάβαση και ε, ε, ε, οι πρόθεσμα οι τυνησιακέ αρχέ θα πρέπει να περιπολούν τι δικέ του ακτέ κατά μήκο τη ακτή, ούτω ώστε οι λαθρέμποροι, οι εγκληματίε, οι δραπέτε να μην μπορέσουν να υποφεληθούν τη έκρηξη κατάσταση. Στη Τινησία επίση είναι να δεχθεί να υποδεχθεί όσου έχουν αποχωρήσει από την Ισία και δεν χρήζουν διεθνού προστασία βάσει τον κανονισμό μα. Για μια πιο διαδρομένη συνεργασία μπορούμε να εξετάσουμε και άλλου στόχου. Παραδείγματο χάρη, πρόθεση προγραμμάτων για να στηρίξουμε το εισόδημα, για να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση στι διάφορε επιμέρου περιοχέ τη νησία, κυρίω για το νότιο κομμάτι τη χώρα. Ευρύτερα, μια συνεκτικότερη προσέγγιση χρειάζεται για πολιτικού ε, ε, για πολιτικούς λόγους, ε, για λόγους οικονομικής ανάπτυξης ε, θα πρέπει να υπάρχουν διατάξεις ούτως ώστε να μπορούν νομίμως να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι υπήκοοι της Τινησίας. Μετά από τις λαϊκές εξεργέσεις διάφορες αραβικές χώρες πιστεύουμε ότι μπορεί να σημειωθούν θετικές εξελίξεις όχι μόνο στην Τινησία αλλά και σε άλλες χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση στη Λαμπεντούζα δεν πρέπει να μειώσει τη βούλησή μας να βοηθήσουμε αυτή την νέα γενιά των αραβικών χωρών που με ειρηνικό τρόπο κατάφεραν να επιτύχουν θεμελιώδεις πολιτικές αλλαγές στο σκηνικό της χώρας τους. Σας ευχαριστούμε κυρία Μάλμστρομ. Τώρα ο κύριος Μπουσουτήλ θα πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατεπίγουσα ανθρωπιστική κατάσταση στην ε, Ιταλία και δει την ίσο της Λαμπεντούζα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κατάσταση η οποία καλεί για κατεπίγουσα δράση. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν πέντε βήματα. Καταρχάς ένα πρόγραμμα τύπου Marshall για την Τινησία και τα άλλα κράτη τη περιοχή, δηλαδή βοήθεια πέραν των σύνορων, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και να αναμένεται η πλήρη συνεργασία των Τινησιακών αρχών ω προ την ε, προστασία των ακτών τους για να αποφύγουμε περαιτέρω τέτοιες ροές ε, λαθρομεταναστών. Δεύτερον, χρειάζεται κατεπίγουσα ανάπτυξη μιας αποστολής ε, της Frontex Rabbits για την ταχεία προστασία των συνόρων. Μια αποστολή Frontex η οποία θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα και να μεταβεί στην περιοχή. Τρίτον, πρέπει να προσφέρουμε στην Ιταλία συγκεκριμένη βοήθεια στην υποδοχή των χιλιάδων αυτών ε, ανθρώπων που έχουν ε, ε, ξοκύλει στη Λαπεντούσα και πρόεδρε δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατό να μας λέτε κυρία Επίτροπε ότι θα αποστείλει η τους ειδικούς της όταν ακόμα αυτή, αυτή η αποκεντρωμένη υπηρεσία δεν έχει ακόμη αρχίσει να λειτουργεί. Πρέπει να βρεθεί κάποια άλλη λύση. Τέταρτο, θα πρέπει να προσφέρουμε βοήθεια στη διαδικασία της επαναπατρισμού άμεσου επαναπατρισμού οποιοδήποτε δεν είναι δικαιούχος προστασίας υπό το καθεστώς του ασύλου ώστε να επιστρέψουν στην Τινησία ή οπουδήποτε προέρχονται. Και πέμπτον θα πρέπει να έχουμε το υπόψη ότι προβλέπεται στη συνθήκη το άρθρο 80, το οποίο ρητά ορίζει πως η πολιτική του ασύλου θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και την, τον ισομερή καταμερισμό των ευθυνών. Είναι νομίζω ώρα πια αυτό το άρθρο να το θέσει σε ορθή εφαρμογή η, συνθήκη, η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπουζούτιλ. Λόμπες Αγγιλάρ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι δεχόμαστε την δημοκρατική, τις δημοκρατικές κινήσεις στις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης. Γνωρίζουμε όμως ότι αυτές οι κινήσεις δεν είναι αυλαβείς. Έχουν επιπτώσεις ως προς τις ε, μεταναστευτικές ροές στις όμορες χώρες. Άρα θα πρέπει να ισχύουν τα άρθρα 67, 77 και 80, διότι θα πρέπει να υπάρχει επιμερισμένη αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση αυτής της ε, πρόκλησης θα πρέπει να πούμε ότι καμία χώρα δεν είναι μόνη της. Δεν είναι θέμα μόνο Ελλάδας, μόνο Ιταλίας ή μόνο Μάλτας. Θα πρέπει να καταδείξουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για, για το Frontex ή την ΕΑΣΟ, αλλά για μια πολιτική απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής διαδικασίας και αυτό που έχει σημασία είναι να δώσουμε μεγάλη σημασία στα κοινά σύνορα και θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της συνολικά. Ευχαριστούμε. Νικολό Ρινάλντι για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, αγαπητέ Επίτροπε, θα ήθελα να σας μιλήσω για την δήλωση του Υπουργών Εξωτερικών της Ιταλίας στη Δαμασκό, όπου είπε ότι η Συρία είναι μια χώρα που ακολουθεί διαδικασίες εξυγχρονισμού ενώ ο Υπουργός μας Εσωτερικών λίγες μέρες ε, πριν απεκδίεται των ευθυνών του και είπε ότι η Ευρώπη θα πρέπει ως συνήθως να αντιμετωπίσει τις ευθύνες της, δηλαδή ως συνήθως αποδίδουμε ευθύνες μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη πως οι αφρικανικές δικτατορίες οι οποίες σήμερα καταβυθίζονται θα ε, τύχουν ενδεχόμενης υποστήριξης. Μιλάμε λοιπόν για 10 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στην Ιταλία το 2009, χρήματα τα οποία δεν χρησιμοποίησε η Ιταλία. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι με αυτές τις δηλώσεις δεν πάει κανείς πουθενά. Δεν κατανοούμε το μάθημα αυτής της εβδομάδας. Η Λαμπεντούζα μας υπενθυμίζει ότι πέρα από τα πολιτικά παιχνίδια και τις πολιτικές δηλώσεις δεν μπορούμε να αγοράσουμε τα πάντα με το χρήμα. Νομίζω ότι κάθε μέρα θα πρέπει η Ευρώπη να μιλά για δικαιώματα και αλληλεγγύη τηρώντας υποχρεώσεις έτσι ώστε να υπάρχει δημοκρατία, ανάπτυξη, τήρηση του διεθνούς δικαίου και ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και καθόλου δημαγωγία. Ευχαριστούμε κύριε Ρινάλντι. Η κυρία Λόχπίλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με τον τίτλο αυτής της συζήτησης υποτίθεται ότι θα προσφερθεί βοήθεια προς την ε, Ιταλία δηλαδή από τα άλλα κράτη-μέλη. Κάνουμε και πάλι το σφάλμα να θέτουμε στο επίκεντρο του προβληματισμού για το άσυλο τα κράτη τα ε, παρόχθια της Μεσογείου. Ενώ θα έπρεπε να θέτουμε τον άνθρωπο και την ανάγκη για προστασία του στο επίκεντρο των συζητήσεων. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζουμε την περίπτωση του κάθε ανθρώπου, σε ποια κατάσταση βρίσκεται και με ποιο τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε τα δικαιώματά του. Δεν θα πρέπει που δεν είναι επιτρέπουμε την επαναπροώθηση των ανθρώπων αυτών και την σφάλιση των συνόρων. Η Frontex δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να είναι χρήσιμη στην κατάσταση. Ενδεχομένως, εάν ε, θέσει το, την προστασία των προσφύγων και τη διάσωσή του στο επίκεντρο των ε, δραστηριοτήτων της, ε, να προσφέρει χρήσιμο έργο. Αλλά μέχρι τότε όχι. Και επίσης η νέα εντολή της Frontex ακόμη δεν έχει κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια πιο διαφανή διαδικασία, καθήκοντα και σύμφωνη με την ε, προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων επιτέλεση του έργου της. Η... Την Ισία βεβαίω θα πρέπει να βοηθηθεί ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της και να είναι και αυτή σε θέση να παραμείνουν στη χώρα τους χωρίς ανησυχία για το μέλλον. Ώστε να προχωρήσει ταχύτατα σε μια οικονομική ανάπτυξη με βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί σε τελευταία ανάλυση αυτή η οικονομική ανάπτυξη και ένα από τα κύρια αιτήματα των ε, ταραχών ε, στην Τινησία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα κράτη αυτά της ε, Μεσογείου στη μοίρα τους δεδομένων των μεγάλων μεταναστευτικών ροών και έτσι είτε πρόκειται για τη Λαμπεντούζα είτε πρόκειται για την Μάλτα δεν θα πρέπει οι εκκλήσεις για βοήθεια να πέσουν σε κοφευόντα ότα. Θα πρέπει να τους στηρίξουμε. Υπάρχουν υποδομές, δυστυχώς όμως δεν υπάρχει πολιτική βούληση και συγκεκριμένη αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λόχπιλερ. Το λόγο έχει ο κύριος Λουί Ταβάρες για ένα Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούμε να συζητήσουμε το πρόβλημα της Λαμπεντούζα ουσιαστικά. Πρωτού ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η νησία του Μπεναλή είχε μία, ένα νόμο που ακόμη δεν ακυρώθηκε, που θεωρεί τη μετανάστευση αξιόπινη πράξη, έγκλημα. Οπότε δεν είναι θέμα Frontex, γιατί ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επιστρέψουν στην ε, φυλακή στην ε, την Ισία και να μεριμνήσουμε για να ακυρωθεί αυτός ο νόμος. Αυτό είναι θεμελιώδες στοιχείο της πολιτικής μας. Δηλαδή πώς εξαρτώμαστε από ένα άτομο, όχι από την κυρία μάλθρομ, ούτε ο κύριος Μπαρόζο. Ο κύριος Καντάφη είναι που επιβάλλει τις εξελίξεις και κανονίζει τι γίνεται με τους μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Επίσης αποδεικνύεται ότι ε, έχουμε 5.000 ακτές ε, έτσι, στον νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και, και πρέπει να προετοιμαστούμε μέχρι... Ε, στην κρίση στην Ουγγαρία δεν είχαμε άλλο προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μαζικές μεταναστευτικές ε, ροές. Ε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει λοιπόν, ε, όπως έγινε με την Ουγγρική Επανάσταση, θα γίνει τώρα με τις λαϊκές επαναστάσεις αραβικές χώρε. θα κάνουμε με αυτές τις μαζικές ροές. Πώ θα υποδεχτούμε του ετούντε άσυλο μέσα στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κύριε Ταβάρες, ο κύριος Βάντερκάμπ ε, θέλει να σας ε, θέσει ένα ερώτημα με τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Δέχεστε το ερώτημα. Όχι. Λάθος χρώμα είδα. Καλά, σας συγχωρούμε. Ας προχωρήσουμε. Κύριος Προβέρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μία άμεση πολιτική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Η ταχεία επέμβαση αφορά ε, στο ότι η Frontex θα πρέπει να έχει μία σαφή διάρθρωση. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει burden sharing, να χρησιμοποιήσουμε τη Europol για ενδεχόμενα τρομοκρατικά στοιχεία κατά τη μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων, καθώς και χρηματικά μέσα για να αντιμετωπίσουμε την έκτακτη κατάσταση. Όμως αυτό δεν επιλύει τα διαρθρωτικά αίτια της επανάστασης του Μαγκρέμπ. Γιατί όπως γνωρίζουμε δεν υπάρχει ελεύθερος τύπος, δεν υπάρχει ελευθερία του συνέρχεσαι και των, του συνέρχεστε και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχουν δηλαδή ε, δημοκρατικά αυτά στοιχεία. Δεν θα μπορέσει λοιπόν να υπάρχει δημοκρατική ανάπτυξη ούτε σταθερότητα σε αυτές τις χώρες. Αυτή είναι η πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Προβέρα. Ο κύριος Μάντλενερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, έχουμε κατάσταση εκτάκτου ανάγκες που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε. Ένα τσουνάμι μεταναστών χτυπάει την Ευρώπη από την Βόρειο Αφρική. Ε, χιλιάδες ετυχοδιώκτες, ακόμη και τρομοκράτες έχουν καταφθάσει στη Λαπεντούσα και εκατοντάδες χιλιάδες ετοιμώσουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Ε, είναι διάτρητα εντελώς τα σύνορα. Και τι κάνει ο Frontex, τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Ε, ε, θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου να οργανώσει βάσει του άρθρου 18.2 έκτακτη σύσκεψη στο Συμβουλίο για να αναλυθούν επίγοντα μέτρα και να αντιμετωπιστεί αυτή η μαζική μεταναστευτική ροή. Ο κύριος, ε, κύριε Μπερλουσκόνη, μη μας ζητάτε λεφτά για τις ε, χωματερές σας, ε, για τους μετανάστες. Σταματήστε να κυνηγάτε τον ποδόγυρο και ασχοληθείτε με τη Βόρεια Αφρική επιτέλους. Ο κύριος Μάουρο τώρα για 1,5 λεπτό από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για τη δέσμευση που έχετε αναλάβει έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατεπίγουσα κατάσταση. Γνωρίζετε πολύ καλά όμως ότι η κατεπίγουσα κατάσταση αποτελεί απόρρια μίας ε, κατάστασης που ζει ολόκληρος ο χώρος του Μαγκρέμπ. Η Ευρώπη είναι ανεπαρκής. Δεν είναι σε θέση να ορίσει μία στρατηγική για τη Μεσόγειο. Πολλές φορές το προσπάθησε, αλλά πάντα απέτυχε. Απέτυχε η διαδικασία της ε, Λισαβόνας ή η διαδικασία ε, συνεργασία της ε, Μεσογείου, των χωρών της Μεσογείου. Σήμερα δεν είναι καν παρόν το Συμβούλιο. Ζητήσαμε από το Συμβούλιο να θέσει το θέμα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για το πρόβλημα όχι τόσο της παράνομης μετανάστευσης, αλλά για το θέμα της δημοκρατίας και της ελευθερίας σε όλο το χώρο της ε, Μεσογείου. Όταν έπεσε το Σοβιετικό μπλοκ, τότε απαντήσαμε συγκεκριμένα με ένα κοινό μέτωπο και δεν λάβαμε υπόψη τους μετανάστες, Πολωνούς μετανάστες που βρίσκονταν ε, στις ε, πατρίδες μας. Κρίναμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική στρατηγική. Χωρίς αυτή τη στρατηγική δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Δηλαδή μιλάμε για καλή θέληση και παραμένουμε εκεί. Ε, θα πρέπει να σας ρωτήσω κατά πόσο μπορείτε να δεχτείτε μια ερώτηση από τον κύριο Πόρτας. Κύριε Πόρτας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε μπορώ να συζητήσω μαζί σας ε, γιατί η Ευρώπη δεν έδωσε απάντηση για όλα αυτά τα προβλήματα, ε, τα μεταναστευτικά. Θα έλεγα λοιπόν, ε, δεν την έδωσε γιατί αστυνομική απάντηση ήθελε να δώσει για ένα οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα. Ε, σας ερωτώ κάτι που σχετίζεται με αυτό που σας είπε και ο κύριος Ταβάρες, ο συνάδελφός μου. Ε, ε, μπορούμε να δεχτούμε ο Frontex ε, και τα επιχειρησιακά του μέσα να χρησιμοποιούνται για τους την ίσιους, ενώ βάσει της οικίας νομοθεσίας προβλέπεται ότι οι μετανάστες φυλακοί θα πάνε ούτως ή άλλως. Χρειάζεται διπλωματική δράση για να κυρωθεί ο νόμος και μετά να αρχίσουμε να συζητάμε άλλου είδους μέσα πέρα από αυτά που προανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Υπενθυμίζω ότι λίγες μέρες πριν με τον συνάδελφο Παντσέρη στην Επιτροπή Μαγκρέπ λάβαμε υπόψη ότι η προσωρινή κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες για να αλλάξει την εσωτερική ένωμη τάξη ως προς το θέμα αυτό. Και επειδή θα πρέπει να υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Ευρώπης και την θα γίνουν προσπάθειες για να επιληθεί το πρόβλημα και σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστούμε κύριε Μάουρο. Υπάρχει κι άλλη μία ερώτηση. Μία ερώτηση προς τον κύριο Ματ Λένερ. Παιδιά... μπαίνε, πρέγω. Ονορεύολε Μέλενκον. Μπορεί να το Μπορείτε να υποβάλλετε το ερώτημα. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Ήταν για τον προηγούμενο μιλητή. Ερωτώ λοιπόν τον συνάδελφο, τι είναι τρόπο απέκτησε την πεποίθηση ότι πρόκειται για Ισλαμιστές και αλίτες ε, όταν μιλάμε για αυτούς τους μετανάστες στη Λαμπεντούζα. Μήπως έχει πέσει θέμα των δικών του φαντασιώσεων ο κύριος συνάδελφος. Πώς το έχει καταλάβει αυτό. Κύριος Ματλενέρ. Ναι, να σας απαντήσω. Εν γέννη, οι άνθρωποι αυτοί που έρχομαι από τη Λιβύη, μουσουλμάνοι, είναι γνωστό, εγκληματίες, ακόμη και τρομοκράτες είναι. Είναι γνωστό τι σπάσει αυτό. Εάν δεν το γνωρίζετε είσαστε αφιλείς. Ωραία, ας προχωρήσουμε. Ο κύριο Σασόλη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε, έχουμε ε, να κάνουμε μια κατάσταση όπου η Επιτροπή αντιμετωπίζει σωστά το ζήτημα, διότι όλοι αυτοί οι μετανάστες δεν βρίσκονται ενώπιον μιας υποδομής, γιατί ότι ε, γινόταν λόγος για μετανάστευση μηδέν πριν ένα χρόνο και έτσι τα κέντρα μετανάστευσης ή συγκέντρωσης είχαν διαλυθεί στη Λαμπεντούζα. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι ιταλικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό. Θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια καταβολής χρημάτων, διότι μιλάμε για συντονισμένες πολιτικές μέσα στα πλαίσια των διεθνών συμβάσεων προστασίας των μεταναστών. Μετά από ορισμένες επικρίσεις που, που ακούστηκαν, θα ήθελα να πω τι, να ρωτήσω τι απαντήσετε όταν η Ιταλική κυβέρνηση ζήτησε την παρέμβαση της Κομισιό. Ο κύριος Μπιτζότο για ένα λεπτό. Λοιπόν από 5.000 μετανάστες έφτασαν στην Ιταλία, ενώ άλλες 100.000 θα μεταβούν προς την Ιταλία, Γαλλία και Γερμανία. Μεταξύ αυτών είχαμε και 11.000 τρομοκράτες ή εγκληματίες. Νομίζω ότι θα πρέπει η Επιτροπή να απαντήσει. Η Βαρόνη Άστον λάμπει δια της απουσίας της. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ανταποκριθείτε. Η σιωπή δείχνει την πραγματική ύπαρξη της Ευρώπης, η οποία φοβάται να αντιμετωπίσει μια κατάσταση τεράστιων ανθρωπιστικών διαστάσεων. Μιλάμε για ιστορικές αλλαγές και επιπτώσεις επί των Ευρωπαίων πολιτών. Τι θα πρέπει να πω στους ψηφοφόρους μου που φοβούνται. Τι θα κάνει αύριο η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτή τη σοβαρότατη κατάσταση. Ευχαριστούμε την κυρία Μπιζότο. Ο κύριος Γιακολίνο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόκειται για ένα πολύ μικρό νησί στο μέσο της Μεσογείου. Ονομάζεται Λαμπεντούζα. Το 2008 έγινε γνωστό αυτό το νησί διότι 40.000 πρόσφυγες βρέθηκαν σε αυτό το μικρό νησί. Όλα αυτά το 2008. Μετά έγινε, συνετάχθη ένα σύμφωνο φιλίας μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης. Η κατάσταση όμως είναι πολύ πιο περίπλοκη. Η νέα κυβέρνηση στην την Ισία και στην Αίγυπτο, οι νέες αυτές κυβερνήσεις, έχουν να κάνουν με αυτές τις ροές. Εγώ είμαι σικελός, αλλά και πολλοί άλλοι μίλησαν για αυτά τα κέντρα αναγνώρισης και έκδοσης. Μιλάμε δηλαδή για αυτά τα κέντρα και μετά το σύμφωνο φιλίας θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει και η Επιτροπή και το Frontex, διότι αυτοί οι ομάδες ταχείας επέμβαση στα σύνορα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Θα θέλαμε το Frontex να αντιμετωπίσει την κατάσταση μαζί με την Λίμπε και τον κύριο Μπουζούτη, να αντιμετωπίσουμε το θέμα το, της χρηματικής αρρωγής. Και ο κύριος Μάουρο ζήτησε από το Συμβούλιο να ε, δράσει άμεσα για να μην χάσουμε χρόνο ως προς αυτή την ε, άμεση προτεραιότητα. Διότι τώρα έρχονται μετανάστες και από την Αίγυπτο και δυστυχώς δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την αξιοπρέπεια αυτών των προσφύγων εξαιτίας αυτών των καθυστερήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, η κυρία Μάλστρομ είμαστε σίγουροι ότι θα δράσει για άλλη μία φορά. Ο κύριος Παντσέρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι μεταναστευτικές ροές αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα ευρωπαϊκών διαστάσεων. Όμως δεν έχει νόημα να εκφράζουμε τη λύπη μας, αλλά να αντιμετωπίσουμε επικοδομητικά και μακροχρόνια αυτό το θέμα. Θα πρέπει να ε, δράσουμε μέσα στα πλαίσια της συνυπευθυνότητας. Θα πρέπει να υπάρχουν τα χρηματικά μέσα για να αντιμετωπίσουμε το όλο ζήτημα και να υπάρχει μία συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την επανακατανομή ευθυνών μεταξύ κρατών μελών. Επίσης θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την προσωρινή κυβέρνηση της Τινησίας για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αναχαιτήσουμε αυτή τη μαζική έξοδο. Είναι αναγκαίο να δούμε εκ νέου την πολιτική γειτονίας θα πρέπει να βασιστούμε σε μια νέα πολιτική οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας και σε μια ευφυή πολιτική μετανάστευσης καθώς και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις μέσα στα πλαίσια της μεταβατικής αυτής πορείας της Τινησίας. Μόνο έτσι θα είμαστε σε θέση να επιλύσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν η Ιταλία και η Ευρώπη. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι αυτή είναι η στιγμή να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Ευχαριστούμε τον κύριο Παντσέρη. Η κυρία Χιμένεθ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κρατώντας αποστάσεις σε θέματα τρομοκρατίας και μετανάστευσης, είδα ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ταχείας επέμβασης όπως την κατάσταση που ζούμε τώρα στη Λαπεντούζα. Είδαμε αυτή τη μαζική έξοδο Ίσιον προς την Ιταλία, που, όπου μιλάμε για μια διαδικασία προαναγγελθέντος θανάτου. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, ε, μη ελεγχόμενη μεταναστευτική ροή. Δηλαδή τι κάνουμε την επόμενη μέρα, ξεχνάμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η στρατηγική της Μεσογείου δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει κοινή πολιτική. Τη στιγμή που δεν συνδράμουμε ε, χρηματικά έτσι ώστε και η Frontex να είναι αποτελεσματική. Νομίζετε ότι η Frontex μπορεί να εγγυηθεί τα ευρωπαϊκά σύνορα. Εγώ νομίζω πως όχι. Ελπίζουμε ότι οι κάτοικοι αυτοί της Τινησίας και της Αιγύπτου κάποια στιγμή να γυρίσουν στη χώρα τους για την ελευθέρωση της οποίας έχουν συνδράμει καταλητικά. Θα πρέπει να προωθήσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική ε, κοινή μεταναστευτικής ε, πολιτικής. Τώρα χρειάζεται περισσότερο από ό,τι ποτέ. Τώρα περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε 17 υποψηφίους ομιλητές. Θα πρέπει να αρκεστείτε στο ένα λεπτό. Η κυρία Αντζελίλη έχει το λόγο πρώτη, η αντιπρόεδρος. Η Ευρώπη είναι η ωραία κοιμωμένη στην περίπτωση των μεταναστευτικών ροών. Σήμερα πληρώνουμε το αντίτιμο. Δυστυχώς δεν αποτελεί η μεταναστευτική πολιτική προτεραιότητα για τα κράτη-μέλη. Αποτελεί μόνο φόρτο για τις όμορες χώρες. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε μια επαρκή στρατηγική ευρωμεσογειακού χαρακτήρα. Δυστυχώς όμως η διαδικασία της Βαρκελόνης δεν απογειώθηκε. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για θέματα που δημιουργούν αμηχανία. Χώρες όπως η Ιταλία, η Μάλτα και η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, ενώ οι άλλες χώρες είναι θεατές, αμέτωχοι θεατές που δίνουν μαθήματα. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει το νομοθετικό έργο και η ενίσχυση των υποδομών. Αναφέρομαι στη Frontex και χρειάζεται και πολιτική θέληση, πρωτίστως. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μάλστρομ και ολόκληρη την Επιτροπή, διότι δεσμεύτηκαν έναντι της Ιταλικής κυβέρνησης για να αντιμετωπίσουμε την έκτακτη κατάσταση της Λαμπεντούζα. Ευχαριστούμε. Πάσκου. Οι γρηταχίε εξελίξει στην Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή πιστεύω έχουν ε, μεταφτρέψει αυτή το ντάουλτσε φαρνιέντε και την αισιοδοξία μα ότι η Ευρώπη δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα και δεν την αντιμετωπίζει καμιά μεγάλη ε, πρόκληση ασφάλεια. Δυστυχώ όμω ε, οι εξελίξει είναι ραγδαίες, ο καιρός, ο χρόνος δεν σταματάει, γι' αυτό κακό συνήθιο και ως εκ τούτου θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και επιτρέψτε μου τώρα να αφαιρθώ στο εξή. Με τις αυξανόμενες ροές μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική κατόπιν των προστατικών εξελίξεων στις περιοχές της χώρας τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να ε, κλείσει τα σύνορά της και τις πύλες της, λέγεται. Εγώ πιστεύω ότι αν θέλουμε να βρούμε μία λύση τεχνολογικού χαρακτήρα πρόβλημα που δεν είναι μόνο χρήματα ή αστυνομική φύλαξη, θα πρέπει να προχωρήσουμε και πέραν των δημόσιων δηλώσεων και αυτές οι δηλώσεις που έχουμε ακούσει από ορισμένου βουλευτές εις βάρος πολιτών κρατών μελών αποτελούν ε, όνειδος και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για όλους μας και όχι μόνο στο ιστορικό αλλά και στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Εκπάσου η κυρία Άλφανο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστούμε διότι ήσασταν διαθέσιμοι άμεσα και σας ευχαριστώ και για τον ε, μελλοντικό, για τον ε, ορίζοντα μάλλον που μας παρουσιάσατε ως προς το θέμα. Υπογραμμίσατε την ανάγκη υποστήριξη της ε, Τινησίας σε αυτή τη δημοκρατική μετάβαση. Αναρωτιέμαι όμως πού πήγαν τα χρήματα που έδωσε η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια στην Τινησία και στη Λιβύη. Σήμερα χαιρετίζουμε αυτή την αφύπνιση των Τινησίων, αλλά γιατί κατασπαταλούσαμε αυτά τα χρήματα τόσα χρόνια. Αν αύριο ε, εγερθούν και οι Λίβοι, τότε θα χάσουμε και τα χρήματα τα οποία θα έχουμε δώσει εκ των προτέρων σε αυτή τη χώρα. Γιατί η Ευρώπη σιώπησε τόσα χρόνια. και μόνο η Αμερική εξέφρασε θέση σε σχέση με αυτά που είπαν οι κύριοι Πόρτας και Ταβάρες μιλήσανε για το γεγονός ότι η μετανάστευση στην Τινησία θεωρείται έγκλημα. Όμως ο, οι μετανάστες ε, τη Λαμπεντούζα που υπενθυμίζει στον κύριο Μάντλενερ ότι δεν προέρχονται από τη Λιβύη αλλά από την, ε, είναι πρόσφυγες διότι σε μία κατάσταση σύγχυσης έπρεπε να φύγουν. Πώς θα τους επαναπατρίσουμε γνωρίζοντας ότι αμέσως θα φυλακιστούν. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την φιλετική πολιτική της Ιταλικής κυβέρνησης που είχε αρνητικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Υπάρχει ένα αίτημα μπλε κάρτας, αλλά δεν ισχύει η διαδικασία κατά το catch the eye. Λυπάμαι. Ο κύριος Μποργέζιου. Εκτός μικροφώνου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την για τη δέσμευση αυτή. Α, αν ε, με όλα αυτά τα χρήματα που δίνουμε και που δίνουμε στους ε, διπλωμάτες, θα, στους διπλωμάτες μας θα έπρεπε να ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβαινε και μην ξεχνάμε ότι στη Σοσιαλιστική Διεθνή συμμετείχε και ο συμπαθής δικτάτορας της Τινησίας με τα γνωστά αποτελέσματα. Θα ήθελα όμως να μας πει η Κομισιόν γιατί δεν μας μιλά σαφώς για την κατανομή που προβλέπεται μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών. Αυτό το ζητούν οι παράκτιες χώρες. Γιατί δηλαδή υπάρχει φόρτος των, των παράκτιων χωρών της Μεσογείου που βρίσκονται κοντά στις χώρες του Μαγκρέμπ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη Frontex. Έσταναν δύο εμπειρογνώμονες στη Λαμπεντούζα ζούμε ένα ανθρωπιστικό δράμα. Δηλαδή, τι, τι κάνετε, ε, στέλνετε δύο εμπειρογνώμονες, χρειάζεται ολόκληρη task force εκεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη βαρύτατη αυτή κατάσταση που μπορεί να επιδεινωθεί και ως προς την κατάσταση της, ε, της υγείας και της υγειονομικής κατάστασης, διότι εκλείπει και το νερό πλέον στη Λαμπετούζα. Επειδή η κυρία Μάλστρομ πρέπει να φύγει στις 6, θα πρέπει να είμαι πολύ ε, αυστηρός με το χρόνο. Για διαφορετικά δεν θα δοθούν απαντήσεις. Ο κύριος Κάσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε, κύριε Επίτροπε, συζητούμε εδώ εδώ και πολλή ώρα αυτή την τραγωδία, μεσογειακή τραγωδία. Και μάλλον δεν προσέξατε αυτά που υπόθηκαν νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει ουσιαστική ελεγγύη στο θέμα της, ε, της ε, μετανάστευσης. Έχουμε μια τραγωδία που εξελίσσεται στη Λαπεντούσα. Έχει κατακλειστεί από μετανάστες στη Λαπεντούσα και όταν πια εξαντληθούν οι δυνατότητες αυτοί όλοι θα μεταναστεύσουν στην ίδια την Ιταλία αλλά Θεός φυλάξει, μην τυχόν και έρθουν στην Μάλτα. Εκεί θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γιατί όποιο έρθει στη Μάλτα, στη Μάλτα θα μείνει. Δεν υπάρχει ε, άλλο, άλλη επικράτεια. Και πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί σε ένα τόσο μικρό νησί. Ούτε να τους εκδώσουμε μπορούμε, ούτε τίποτε άλλο. Χρειαζόμαστε λοιπόν δέσμευση από τα άλλα κράτη, κυρίως από τα κράτη της Βόρειας Ευρώπης. Όπω είπε πολύ σωστά και ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, αυτή την αλληλεγγύη δεν τη βλέπουμε από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κροτσέτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο διότι προσέδωσε τη σωστή σημασία στο θέμα της θυνησίας και θα ήθελα να, μιλήσουμε, να μιλήσουμε για υποστήριξη της θυνησίας και των άλλων χωρών που καταπολεμούν τις δικτατορίες και κινούνται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως ε, μία από τις μεγαλύτερες ε, δυνάμεις, η Ιταλία, αντιμετωπίζει πρόβλημα για το πώς θα υποδεχτεί 5.000 πρόσφυγες στη Λαμπεντούζα. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το πορθμίο προς τη Σικελία που κινείται κάθε μέρα και μπορούμε να τους ε, μεταφέρουμε και προς το αεροδρόμιο. Όμως αυτή τη στιγμή δεν ε, μιλάμε το, για το θέμα του Frontex και για το πώς θα σταματήσουμε τις αποβάσεις. Έχουμε να κάνουμε με χώρες και με πολίτες που τάσσονται υπέρ ενός δημοκρατικού καθεστώτος. Τώρα όμως έχουμε τη δυνατότητα να τους ε, υποδεχτούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να επεκτείνουμε τους ορίζοντές μας και να τους χορηγήσουμε ακόμα και θεωρήσεις. Μόλσερ. Κύριε Πρόεδρε, μαζικές ροές προσφύγων όπως αυτές που βλέπουμε τώρα ε, από την Τινησία. Είδαμε το 89 ίσως με την κατάρρευση του κομμουνισμού όπου πάλι δεν είχε προβλέψει αυτές τις εξελίξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατελήφθη εξαπίνης. Το ίδιο και τώρα. Και καλείται η Ιταλία να μην επαναπροωθήσει αυτούς τους πρόσφυγες από την Ισία. Αυτό όμως είναι ακριβώς το πρόβλημα, ότι αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν επαναπροωθηθούν με κάποια βοήθεια για την ε, πάνωδο στην πατρίδα τους, θα πρέπει να διοχετευτούν κάπου αλλού. Έχουμε να κάνουμε με ετούντες ε, το άσυλο οι οποίοι έχουν ε, μια κάποια οικονομική επιφάνεια πολλές φορές και που με τη στάση αυτή διονγκώνουν το φαινόμενο της ε, μετανάστευσης και των προσφύγων. Πρέπει να σχεδιάσουμε διαφορετικά την πολιτική μας. Ευχαριστώ πολύ Σιλβέστρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστούμε που τουλάχιστον μας ε, τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ για όσα είπατε, για τις δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει και αποδεικνύει πώς ένα συντονισμός μεταξύ Ευρώπης και Ιταλίας μπορεί να βοηθήσει τη χώρα μου να αντιμετωπίσει την κατεπίγουσα αυτή ανάγκη. Επαναλαμβάνω μιας φράσης Υπάρχει ένας νέος άνεμος που φύσα στην ε, κεντρική, Αμερική, κεντρική Ευρώπη, όπως είπατε. Είναι όντως ελευθερία και δημοκρατία που δίνει τις άμεσες επιπτώσεις και που πρέπει να διαχειριστεί τώρα η Ιταλία. Εάν δυναμώσει ο άνεμος, συμβαίνει, να συμβαίνει να μα πέφτουν οι πύργοι τους οποίους ε, έχουμε φτιάξει πάνω στην άμμο. Στην Πούλια, στην Νότιο Ιταλία από προερχόμαστε, είναι εκατοντάδες που κατασκευάζουν πύργους, δηλαδή μορφές ε, φιλοξενίες που δεσμεύονται και που δίνουν για να εγγυηθούν αξιοπρεπή υποδοχή των μεταναστών. Μόνοι μας όμως δεν τα καταφέρνουμε. Καλό θα ήταν, κυρία Επίτροπε, αν αυτοί οι πύργοι που εδώ και χρόνια κατασκευάζουμε να έχουν και ένα σήμα και να σηματοδοτούν και μια Ευρώπη, η οποία βοηθάει και προσέχει. Ευχαριστούμε. Κύριε Σμούλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μοιάζει λίγο ηρωνικό τώρα που ανακοινώνεται ελευθερία και δημοκρατία στην Τινησία να ξεκινάει ένα κύμα προσφύγων. Και τώρα ακριβώς εγκαταλείπουν αυτοί οι άνθρωποι τη χώρα. Λίγο δυσνόητο μου φαίνεται. Ίσως λοιπόν να έχουμε εδώ πέρα ένα προμήνυμα του τι έρχεται. Καλό είναι λοιπόν η Κομισιόν να προετοιμαστεί με όλα τα δυνατά μέσα και τώρα θα πρέπει να αποδείξει η Κομισιόν πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Όλα τα κοινοτικά μέσα θα πρέπει να λειτουργήσουν, θα πρέπει να βοηθήσουμε την Τινησία, αλλά μου φαίνεται αναπόφευκτο πως σε αυτή την περίπτωση ακριβώς τώρα που ανακοινώνεται η ελευθερία στην Τινησία να έρχονται άνθρωποι οι οποίοι μάλλον δεν μου φαίνονται να είναι πραγματικοί πρόσφυγες. Γι' αυτό θα πρέπει η Κομισιόν να δει πώς θα μπορέσουν να επαναπροωθηθούν αυτοί οι άνθρωποι στην Τινησία για να στείλουμε ακριβώς το παράδειγμα που πρέπει. Ευχαριστώ κύριε Μόλτερ, κύριε Σφιντάντσα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η φοβερή και έκτακτη εισρωή των μεταναστών που φτάνουν στι νότιε ακτέ Ιταλία αναγνωρίζει την μεγάλη επιτάχυνση. Πρέπει να υπάρχει επιτέλου μια κοινή προσέγγιση στη διαχείριση του φαινομένου αυτού. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, να εξελίξει διάλογο μεταξύ Ιταλικών Αρχών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά με θετικό τρόπο, με στόχο να δοθεί μια απάντηση στην κατεπίγουσα ανθρωπιστική ανάγκη που αντιμετωπίζουμε. Μπορώ να πω, συμφωνώντα με τον συνάδελφο το θέμα δεν είναι τόσο οι 5.000 που έχουν φτάσει μέχρι στιγμή, αλλά η διάσταση ενδυνάμει τεράστια σε, σε διαστάσει αποκάλυψη. Χιλιάδε μπορούν να φτάσουν ακόμα στι ακτέ μα, εάν δεν στείλουμε συγκεκριμένα πολιτικά μηνύματα. Και πρέπει να δεσμευτούμε προ αυτή την κατεύθυνση με όρου πραγματικά του κατεπήγοντο. Το κατεπήγον πραγματικά θα, θα ξεπεραστεί, αλλά πρέπει να δώσουμε μια πραγματικά δομημένη διδαχτική λύση. Να δημιουργήσουμε κάποιε συνθήκε άμεση διαχείριση των διαδικασιών αυτών. Εντοπισμού, επαλήθευση του καθεστώτο των μεταναστών, των προσφύγων και ενδυνάμει του επαναπρόθεσή του. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τι ε, υπηρεσίε Interpol για να εντοπίσουμε ενδεχόμενα κλιματικά στοιχεία στα μεταναστευτικά αυτά ρεύματα. Νομίζω ότι έχει σωστά απαντήσει το, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο από κοινού. Ευχαριστούμε. Κυρία Ρομέρο Ρόπελ Κάρμεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω το εξή από την κυρία Επίτροπο, γιατί ξέρετε πως ε, αυτό το απόγευμα ακουστήκαμε ίσως και λίγο ιστερική σε αυτό που είπαμε. Πείτε μου, αυτοί οι 5.000 που φτάσανε στη Λαμπεντούσα είναι τρομοκράτες. Δεν μπορούμε αυτό να το αποδείξουμε. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Έχουμε, νομίζω, αρκετούς μηχανισμούς αντικατασκοπίας και δυνάμεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να μας εξηγήσουν τι άνθρωποι είναι αυτοί γιατί αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που φτάνουν με τις αυτοσχέδιες βάρκες ίσως θα έπρεπε αντί να τους θεωρούμε τρομοκράτες να πάμε να τους επισκεφθούμε και να δούμε ακριβώς ε, πώς ε, ζουν και καλό θα ήταν να πάμε και στην Τινησία μια επίσκεψη γιατί ίσως αυτοί που έφτασαν ε, στην Λαμπεντούσα ήταν από το ιστορικό της χώρας, από τις ζώνες εξόριξης μετάλλων, όπου ζουν σε συνθήκες απίστευτες φτώχειας και καταπίεσης από τους ε, από το καθεστώς Μπεναλή. Λοιπόν, πριν τους αποκαλούμε τρομοκράτες, παρακαλώ ας δούμε ακριβώς ποιοι είναι. Κυρία Φαζόν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, μια νέα ανθρωπιστική τραγωδία λαμβάνει η χώρα στο κατόφλι της Ευρώπης η Λαμπεντούζα σήμερα και ίσως να έχουμε αύριο ακόμα μεγαλύτερη ροή ανθρώπων από τις άλλες χώρες. Από την Αίγυπτο μόνο έχουμε 600 άτομα κάθε μήνα και δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Χρειάζεται μια γρήγορη κοινή απάντηση. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι να κλείσουμε την πόρτα και η απάντηση δεν μπορεί να, ε, τους εξισ... να είναι να τους εξισώνουμε με τους ε, τρομοκράτες. Ε, η Ευρώπη έχει μια θεμελιώδη ελευθερία που είναι η ελευθερία διακίνησης των ανθρώπων, οπότε δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε με τέτοιου ανθρώπου. Πρέπει να μοιραστούμε το βάρο αυτό, να μοιραστούμε οικονομικού και άλλου πόρου. Μιλάμε για ανθρώπινε ζωέ εδώ πέρα, οι οποίε κινδυνεύουν. Η απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα γεγονότα στην Αίγυπτο δεν ήταν αυτή η οποία έπρεπε. Πρέπει να μην έχουμε επίσης ε, ξενοχωρικές αντιμετωπίσεις από διάφορα κόμματα. Η Ιταλία χρειάζεται βοήθεια τώρα και πρέπει να τη δώσουμε το στο μοντρινατόν. Φάνονται κάποια ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θετικές οι δημοκρατικές εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική, αλλά βεβαίω αυτό σημαίνει κάποιε υποχρεώσει για την Ευρώπη και τα προβλήματα της ε, Βορείου Αφρικής δεν μπορούν να λυθούν στη Νότια Ευρώπη. Οπότε εδώ πέρα είμαι αλληλέγγυος με τους Ιταλούς συναδέλφους. Αλλά το ερώτημα προς ε, την Επίτροπο είναι ποιες είναι οι δυνατότητες για να γίνουν πιο γρήγορες οι διαδικασίες, να κρυθούν πιο γρήγορα αυτοί οι άνθρωποι και να τους αποστείλουμε αν δεν είναι πρόσφυγες πίσω στην Τινησία γρήγορα. Γιατί βλέπουμε τώρα μεγάλες ομάδες νέων ανδρών που πάνε προς την Νότια Ιταλία θα είναι από αυτούς πολύ οικονομικοί μετανάστες και πρέπει να ξεχωρίσουμε τους πραγματικούς πρόσφυγες από τους οικονομικούς πρόσφυγες. Και μετά υπάρχει το ζήτημα της επικοινωνίας. Πολλοί Ευρωπαίοι θεωρούν πως πολλοί την ίση πάνε στη Νότια Ιταλία. Αυτό είναι πρόβλημα επικοινωνίας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε επιταχύνεται τις διαδικασίες και καλύτερη επικοινωνία. Η κυρία Ήρς, παρακαλώ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ήμασταν ε, όλοι ικανοποιημένοι, χάρη και το κοινό για την επανάσταση στην ε, την Ισία και την Αίγυπτο ε, και τώρα πλέον υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία στην ημερήσια διάταξη. Και τις τελευταίες μέρες αυτό κυριάρχησε. Όμως εδώ και δύο-τρεις ημέρες κυριαρχούν οι εικόνες των ροών προσφύγων, ανθρώπων σε βάρκες. Αυτά γεμίζουν τα ΜΜΕ και τις εφημερίδες. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα έτσι ώστε τελικά να μην χάσουμε αυτή την αποφασιστική στιγμή και να μείνουν μόνο οι εικόνες προσφύγων αλλά να δούμε και το τι έχουν επιτύχει αυτές οι χώρες. Και αυτό πρέπει να το πούμε στο κοινό, πως έρχονται τώρα πολλοί άνθρωποι, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ανθρώπων θα επιστρέψει, γιατί δεν έχει δικαίωμα ασύλου στις χώρες μας. Οπότε πρέπει να τεθεί και το ερώτημα των οικονομικών προσφύγων. Και σαφές είναι και το εξής, εάν αυτοί οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν προοπτική, θα επιστρέψουν ξανά και ξανά και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα κάποτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαλαβράκος έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η Μεσόγειος λέγεται, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι αντιληπτό λοιπόν ότι οι μεταναστευτικές ροές θα διευρυνθούν. Ε, πρέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους αντιμετωπίζουμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι, σαν ανθρώπους. Βεβαίως όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι το μέγα πλήθος των μεταναστών προέρχεται από μουσουλμανικούς πληθυσμούς. σύμφωνα με την επίσημη έκθεση οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην εικοσαετία που έρχεται θα αυξηθούν κατά 35% και από 1,6 δις θα φτάσουν σε 2,2 δις. η ευρώπη σήμερα έχει μόλις 2,7 των κατοίκων της μουσουλμάνους αναμένεται με αυτές τις ροές και με αυτές τις γεννήσεις να φτάσει στο 20 χρόνια μετά να έχει περί το 6%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι επέρχεται μια οικονομική και κοινωνική ανατροπή στη λειτουργία της Ευρώπης, στην κουλτούρα της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να το δούμε το θέμα σαν Ευρώπη και να μην αφήνουμε τα κράτη-μέλη να το αντιμετωπίζουν μόνοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε η επίτροπο, η άνεμη τη αλλαγή πνέουν ε, ισχυρά από την Βόρεια Αφρική και κάπως μα θυμίζει ότι είχε συμβεί στην Ανατολική Ευρώπη πριν από 20 χρόνια. Εάν το αποτέλεσμα κατά πότε είναι το ίδιο, πλέον πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με εγκαθίδρυση δημοκρατικών, ε, επανα, ε, εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτευμάτων. Ταυτόχρονα όμω το αρνητικό είναι ότι έχουμε και μεγάλα ναυτικά ρεύματα. Τεράστιο πρόβλημα στην Νότια Ιταλία με τι εισρωέ, αλλά, και, ευρύτερα την Ευρώπη. Άρα η λύση πρέπει να είναι ευρύτερα ευρωπαϊκή. Δεν μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα στου ε, πρόσφυγε, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούν να ανοίξουν διάπλατα οι θύρε σε όλου ανεξαιρέτω πρόσφυγε. Η λύση λοιπόν θα έγκυται νομίζω σε ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα και πολιετέ, όπω πρότεινε η συνάδελφο κ. Μπούσετιν, ώστε ο επαναπατρισμό να λαμβάνει χώρα όταν θα πρέπει, με ασφαλή και σωστό τρόπο, και ταυτόχρονα να δοθεί δυνατότητα ε, σε αυτού οι οποίοι ε, ζητούν άσυλο αλλά που δεν έχουν το δικαίωμα να επαναπροωθηθούν. Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη για να το κράξουμε. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε είναι πανευρωπαϊκό. Η Ευρώπη πρέπει να δείξει άλλη αλληλεγγύη και να εμφανιστεί ενωμένη. Τώρα έχουμε προβλήματα με τους πρόσφυγες από την Τινησία στην Ιταλία, αλλά μπορούν να προσθούν και άλλες χώρες, η Λιβύη, η Αίγυπτος και ήδη σήμερα έρχονται χιλιάδες άνθρωποι από αυτές τις ε, χώρες και μπορεί να αυξηθούν αυτά τα ρεύματα ακόμα. Εάν ε, το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρω τι θα γίνει. Και λυπούμε για το ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Πρέπει να τα συζητήσουμε με το Συμβουλίο και με την Κομισιόν να βρούμε καλές ε, νομικές ορθά λύσεις και όπως υπόθηκε δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους τους πρόσφυγες εδώ πέρα της Βορείου Αφρικής. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Αυτοί οι οποίοι δεν ε, μπορούν να λάβουν πολιτικό άσυλο πρέπει να επιστρέψουν στις χώρες τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουμουτσάκος θα τελειώσει ε, την συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, καλώς ορίσατε σε αυτή την συνάντηση. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Σήμερα το πρόβλημα είναι στη Λαμπεντούζα. Αύριο θα είναι στη Μάλτα και στην Κρήτη μεθαύριο και ας μην γελιόμαστε θα είναι στο μιλάνο μετά από λίγο θα είναι στις βρυξέλλες θα είναι στο παρίσι. το πρόβλημα δεν είναι των χωρών εταίρων του νότου είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. απαιτείται αλληλεγγύη. απαιτείται επίση να ενισχύσουμε τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μα και τα μέσα είτε frontex europol θαλάσσια επιτήρηση. αλλά επίση, κυρία επίτροπε είναι πολύ σημαντικό 8 χρόνια μετά την θέση τους εφαρμογή να ξαναδούμε σοβαρά και να αναθεωρήσουμε όπου χρειάζεται τη συμφωνία δουβλίνο 2. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, κλείνω, γιατί έχει ήδη λάβει χώρα μια ώρα συζήτηση. Λυπάμαι, κλείνει ο κατάλογος αγορετών. Δίνω το λόγο στην κυρία Επίτροπο για να κλείσει όλη η συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση αυτή. Αν είχε ακούσει ο κ. Μπουζούτη τι είχα πει στην εισαγωγή μου, θα είχατε ακούσει ότι είπα σχεδόν τα πάντα που περιλάβατε στην ομιλία σας, αλλά ευχαριστώ να τα επαναλάβω. Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα, ώστε να βοηθήσουμε άμεσα τι αλληλικέ αρχέ. Είμαστε σε διάλογο μαζί του για να δούμε τι ακριβώ βοήθεια χρειάζονται. Η Ιταλία έχει πολύ μακρά εμπειρία στην αντιμετώπιση διαφόρων, ε, διαφόρου τύπου καταστροφέ, αλλά ίσως σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια για τα θέματα παροχής καταφυγίου, για φάρμακα, για ψηφιστική βοήθεια και ίσως βοήθεια για μια έλεγχο, ε, ταυτοποίηση την αναζήτηση του άσυλο κλπ. Ναι, όντω είναι ευρωπαϊκή ευθύνη και γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε ευρωπαϊκέ λύσει. Έχουμε προσωπικό του Frontex επιτόπου, αλλά επίση εξετάζουμε την δυνατότητα, την πιθανότητα και ήδη είμαστε έτοιμοι να στείλουμε σχετικό κλιμάκιο Frontex άμεσα. Αλλά πρώτα πρέπει να συζητήσουμε του τρόπου και τη διαδικασία με την Ιταλία, αλλά και με άλλε χώρε που ενδεχομένω μπορούν να συνεισφέρουν και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριο Μπιζουτελή ε, είναι ο εισηγητή για τη Frontex. Οπότε στο μέλλον ελπίζω ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερη λειτουργία του οργάνου αυτού με τι τροποποίησει που θα γίνουν. Εάν έχουμε επιχειρήσει σε ύδατα τη Τινησία Frontex, προφανώ πρέπει να το κάνουμε πάλι σε συνεργασία με τι Τινησιακέ Αρχέ. Αλλά δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Ενθαρρύνουμε επίση τι Τινησιακέ Αρχέ να να δεχθούν και πάλι πίσω τους ε, υπηκόους τους που δεν χρήζουν διεθνούς βοήθειας. Εξετάζουμε το νόμο αυτό που το θέμα που έθιξε ο κ. Σταβάρας και άλλοι. Ελπίζουμε ότι η δημοκρατική κυβέρνηση να μην έχει τέτοιου είδους νόμο, αλλά βέβαια πρέπει να εξεταστεί κατά περίπτωση και να τον εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Επίση, είμαστε πρόθυμοι να υποστηρίξουμε τι συνεχιακέ αρχέ με συμβουλευτικέ υπηρεσίε, ε, με την δημιουργία περιπολιών και διασυνοριακών περιπολιών και επίση με σχετικά κονδύλια. Και επίση, υπάρχει και μια σχετική λειτουργία ε, και στην ε, Μάλτα και μπορούν να στείλουν σχετικά κλιμάκια αν χρειαστεί. Στην επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα ζητήσω το θέμα που πρόκειται να συνέλθει και επίσης εργαζόμαστε με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για να τους ζητήσουμε επίσης να βοηθήσουν, για τους πρόσφυγες να μας, βοηθήσουν επίσης για να συζητήσουμε το σχετικό θέμα και να μας βοηθήσουν να κάνουμε μια σχετική ανάλυση για το μέλλον. Frontex επίσης εμπλέκεται στην εκπόνηση μιας ανάλυσης για την ευρύτερη περιοχή. Στην Δινησία, όπως περισσότερο είπατε, είναι μια θετική και επίφορη, να θέλετε, ε, ελπιδοφόρα κατάσταση και όλοι υποστηρίζουμε μια δημοκρατική μετάβαση. Η Lady Άνστον ήταν σήμερα εκεί να συζητήσει. Προσφερθήκαμε να παράσχουμε βοήθεια στις προβλεπόμενες εκλογές. Συζητούμε διαφορετικούς τρόπους για την ενίσχυση και διαφορετικού τύπου αρρωγής για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη δημοκρατικών θεσμών. Η οικονομική αρρωγή επίσης μπορεί να παρασχεθεί. Συζητούμε διάφορα προγράμματα κινητικότητα και πρέπει να επαυξήσουμε τη δυνατότητα ανθρώπων να έρχονται νομίμω στην Ευρώπη και βέβαια ε, θα υπάρξει και σχετική συζήτηση στην διάσκεψη Ντόνα. Βέβαια, συμφωνώ ότι πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο τη περιοχή. Πολλοί θα εκπλαγούν. Πολύ εξεπλάγημεν όταν έπεσε το τείχο του Βερολίνου. Δεν είχαμε ένα άτομο πρόγραμμα δράση. Η κατάσταση μπορεί να είναι λίγο διαφορετική τώρα, αλλά βέβαια ότι οι άνθρωποι ζητούν ελευθερίε και δημοκρατία είναι κάτι το οποίο πρέπει να υποστηρίξουμε εμεί στην Ευρώπη. Βλέπουμε το σχετικό όλο σχέδιο πολιτικό και στις γειτονικέ μας χώρες γιατί οι συγκυρίες το απαιτούν και βλέπουμε ευρύτερα την περιοχή και την Αίγυπτο αλλά και την ευρύτερη περιοχή πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα διάφορα εργαλεία, τους μηχανισμούς, τα ταμεία και πολιτικές που έχουν στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να τα διαμορφώσουμε επακριβώς και να, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαφαινόμενε συνθήκες, νέες συνθήκες στην αγορά, στην περιοχή, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ε, για τη συζήτηση. Το θέμα ήρθε στην μέση διάταξη και πιθανότητα θα παραμείνει στην επικαιρότητα για πολύ διάστημα. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή ε, παρακολουθεί εκ του σύνεγγης ε, την κατάσταση και προτίθεται να βοηθήσει και την Ιταλία και την Τινησία και σε άλλες χώρες όπως προκύπτει. Ευχαριστούμε κυρία Μάλστρομ και με την παρέμβασή σας ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτή και τώρα στην ημερήσια διάταξη περάμε στην έκθεση της κυρίας ε, Όμεν Χόιτεν πάλι στα θέματα των ε, επαρκών βιώσιμων και ασφαλών ευρωπαϊκών συνταξιδιωτικών συστημάτων στην Ευρώπη. Δίνω λίγο χρόνο για να αλλάξουν θέσεις οι επίτροποι. Ψάχνουμε την κυρία Σιγή.